Περίεργη μετάφραση, αλλά δεν ξέρω αν το κατάλαβε. die επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση τα πρακτικά της χθεσινή συνεδρίασης και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι στην διάθεσή σας υπάρχουν αντιρρήσεις δεν βλέπω κάποια αντίρρηση άρα τα πρακτικά εγκρίνονται Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει καθυστερήσει λίγο γιατί βρίσκεται ακόμα στην συνεδρίαση της ε, Αρμόδιας Επιτροπής οπότε θα ε, μιλήσει λίγο αργότερα και τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Thank you so ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να εκφράσω καταρχάς προσωπικά μου συλληπιτήρες οικογένειες και στους φίλους των εκατοντάδων θυμάτων στη Μοζαμβίκη, στο Μαλάουι και στη Ζιμπάμπουε οι σκέψεις μας είναι με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επλήγησαν από αυτή την καταστροφή. Επανειλημμένα έχω πει σε αυτή την αίθουσα ότι η Ευρώπη σημαίνει αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη όχι μόνο εντός Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής. Στεκόμαστε στο πλευρό και των τριών χωρών με κατεπίγουσα χρηματοδότηση, με ενίσχυση σε είδο και εμπειρογνώμονε επίση που μεταβαίνουν επί τόπου. Να συνοψίσω ποια είναι η ευρωπαϊκή ανταπόκριση σε αυτή την καταστροφή. Καταρχάς χρηματοδότηση. Λίγες ώρες μετά την άφηξη του κυκλώνα σε αυτές τις περιοχές απελευθερώσαμε ένα πακέτο βοηθείας ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για να διευκολύνουμε την πρόσβαση με αεροπορικέ συγκοινωνίε και να πλησιάσουμε αποκλεισμένε περιοχέ και κοινότητε για να του δώσουμε στέγαση, νερό και υγειονομική περίθαλψη. Στι 9 Απριλίου κινητοποίησαμε πέραν αυτών άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τις τρεις χώρες, για στέγαση, για νερό, τρόφιμα, υγεία ε, και κοινωνική υποστήριξη. Οπότε η συνολική βοήθεια φτάνει σε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση σε είδο μέσω 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήσεων αναπτύξαμε μέσω του Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προστασία των Πολιτών διάφορα είδη ανακούφισης των πληγέντων που έχουν προσφερθεί από εννέα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, του Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Δανία. Προσεφέρθησαν αυτά τα είδη. Είμαι ευγνώμων προ αυτέ τι χώρε. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε 57 χάρτες Κοπέρνικος και χορηγήσαμε τις χάρτες στη Μοζαμβίκη, το Ζιμπάμπουε και στο Μαλάβι τους χάρτες αυτούς, τους δορυφορικούς. Μετά για τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων. Εκεί στείλαμε οκτώ ειδικού για ιδεολογία και επιδημιολογία επιτόπου για να κάνουν αξιολόγηση και να βρουν την κατάλληλη απάντηση στα προβλήματα των τριών χωρών και να αντιμετωπιστεί και ε, τα, η επιδημία χολέρας που ξέσπασε πρόσφατα. Και μια ομάδα πολιτικής προστασίας 13 μελών που μετέβη στις 23 Μαρτίου μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πήγαν εκεί και θέλουμε να στείλουμε και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη μας. Όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες είναι στη Μοζαμβίκη τώρα που μιλάμε και βοηθάνε, σώζουν ζωής, ζωές συγγνώμη επιτόπου να κατονομάσω αυτές τις ομάδες, διότι πιστεύω ότι πρέπει να τους δείξουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι οι ομάδες μας μπορούν να κάνουν έξοχη δουλειά επί τόπου. Όπως σας είπα, είναι ακόμα στη Μοζαμβίκη αυτοί οι άνθρωποι, διότι είναι πραγματικά ήρωες εκεί. Πορτογαλία. Έστειλε μια ομάδα έρευνας και διάσωσης, μια τρική ομάδα, το Λουξεμβούργο, ομάδα